και σίγουρα οι αποφάσεις ε, και οι λύσεις που εφαρμόζονται σε χώρες υψηλού εισοδήματος δεν πρέπει αναγκαστικά να ακολουθηθούν και σίγουρα δεν πρέπει να επιβληθούν και στα άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έλξε εδώ <clears throat> και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι δήλωση της Επιτροπής με θέμα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης στις υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον επίτροπο τον κύριο oettinger εξ ονόματος της επιτροπής. Η 20 Απριλίου ήταν ε, μαύρη μέρα για τον κόλπο του Μεξικού, για τις Ηνωμένε Πολιτείες, για τον κόσμο ολόκληρο. Πριν από τέσσερις ακριβώς εβδομάδες, η βιομηχανία και οι κρατικές αρχές καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες μέχρι τώρα άκαρπες για να σταματήσουν την τεράστια διαρροή πετρελαίου και να ε, μειώσουν τις περιβαλλοντικές ε, επιπτώσεις. Βλέπουμε από το ατύχημα αυτό πώς οι κίνδυνοι συνδέονται με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και τις θαλάσσιες εξέδρες. Σωστά αυξήθηκε η συνειδητοποίηση του κόσμου, όχι μόνο στι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Νορβηγία παράγει πάνω από 200 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου το χρόνο. Από τη Βόρεια Θάλασσα τον περισσότερο. Οι εξορίξεις και οι ε, ερευνητικές ε, ε, προσπάθειες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο βέβαια διαφέρουν γιατί δεν είναι τόσο βαθιά όσο στο κόλπο του Μεξικού. Θα πρέπει και εμείς να προσέχουμε να δούμε τι θα γίνει σε περίπτωση ατυχήματος και να εξοπλιστούμε κατάλληλα για να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό έχουμε αρμόδια όργανα και μηχανισμούς έτσι ώστε γρήγορα να μπορούμε να αντιδρούμε σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στην Αυσιπλοεία. Έχουμε και ε, μηχανισμούς προστασίας, ε, πολιτικής προστασίας και ε, σκάφη, καλή συνεργασία και συντονισμό. Και η συνάδελφος Γεωργίευα ακριβώς ήδη από νωρίς ενέκρινε και, και μάλιστα πρότεινε ευρωπαϊκή βοήθεια και για τον κόλπο του Μεξικού. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η πρόληψη για να μην χρειάζεται να δρούμε εκ των υστέρων μετά από μια τόσο μεγάλη καταστροφή. Με τον συνάδελφο Επίτροπο κύριο Ποτότσνικ παρακαλέσαμε από κοινού τις υπηρεσίες να κοιτάξουν την ομοθεσία μας ε, στον τομέα αυτό και να την ελέγξουν ε, για να είναι ένα πλαίσιο προστασίας ε, και του περιβάλλοντος και σε γενικές περιπτώσεις και σε ειδικές, σε συγκεκριμένο ατύχημα. Οι οδηγίες μας ε, χρειάζονται ε, προδιαγραφές ελάχιστες για τον εξοπλισμό και ε, αναφέρουν και λεπτομερείς προδιαγραφές για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων. Ε, όλα λοιπόν αυτά τα νομοθετήματα που έχουμε θα πρέπει να τα ελέγξουμε, να τα επαληθεύσουμε αν είναι επαρκή για τη χειρότερη περίπτωση, για ένα τέτοιο σενάριο καταστροφικό. Και εδώ χρειάζεται στενή συνεργασία και με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές γιατί ένα μεγάλο τμήμα των ορισμών ασφαλείας και των διατάξεων ασφαλείας είναι στα χέρια των κρατών μελών μας και όχι άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, καλή η νόμη, αλλά δεν είναι 100% εγγύηση. Πολλά θα εξαρτηθούν από ε, τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις ε, και τη δράση και λειτουργία της βιομηχανίας μας. Γι' αυτό έχουμε κάθε λόγο να συνεργαζόμαστε. Η πολιτική και η οικονομία θα πρέπει να συνεργάζονται για να βεβαιωθούμε ότι το περιβάλλον και η κοινή ε, γνώμη είναι όσο γίνεται πιο ασφαλής. Η ε, ασφάλεια θα πρέπει επίσης να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων που έχουμε με φορείς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Γι' αυτό την περασμένη εβδομάδα συγκάλεσα ένα μεγάλο ε, όργανο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και ήταν και η κυρία Γεωργίευα, η συνάδελφος παρούσα. Σε αυτή τη συνεδρίαση λοιπόν που ήταν στραμμένη ακριβώς αυτό το αντικείμενο, καλέσαμε τη βιομηχανία να εξασφαλίσει ότι καταλαμβάνει αναλαμβάνει συγγνώμη κάθε ε, προσπάθεια, κάθε πρωτοβουλία για να αποφευθεί ε, ένα παρόμοιο επεισόδιο. Ε, δώσαμε ένα ερωτηματολόγιο και καλούνται οι εταιρείε να απαντήσουν πολύ συγκεκριμένα τις επόμενες ημέρες τι κάνουν για την ασφάλεια στις εξέδρες εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και ε, τι κάνουν για να προστατεύουν τα ύδατα και τις ακτές των κρατών μελών. Αυτή τη συνάντηση λοιπόν με τον κλάδο τη θεωρώ στην αφετηρία και την αρχή μια διαδικασία ολόκληρη που ενισχύει τη διαφάνεια του τρόπου λειτουργία των εταιριών αυτών για να δούμε πόσο τηρούν τι προδιαγραφέ και πώς ε, εφαρμόζουν τι καλύτερε τεχνικέ. Προγραμματίζουμε του επόμενου μήνε και δεύτερη συνεδρίαση όταν θα έχουμε καλύτερη αντίληψη, καλύτερη εικόνα για ε, τις ε, καταστάσει και όταν θα έχουμε βγάλει τα διδάγματα από τον κόρπο του Μεξικού. Αυτή τη στιγμή αναλύουμε ακόμα ε, τις καταστάσεις και τα αίτια. Θα ήταν πολύ ε, πρόωρο να βγάλουμε νέα συμπεράσματα ή να ζητήσουμε νέα νομοθεσία. Αν όμως διαπιστωθεί ότι χρειάζεται αλλαγή της νομοθεσίας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα διστάσει να κάνει προτάσεις για ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Βλέπετε λοιπόν κυρίες και κύριοι βουλευτές ότι στην Ευρώπη ε, συνεχώς κάνουμε προσπάθειες να αποφύγουμε ε, αντίστοιχη τραγωδία ε, στα δικά μας ύδατα. Αν συμβεί όμως το απευκταίο, έχουμε πολλά μέτρα και μηχανισμούς και χωρίς καθυστέρηση θα μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά για να προστατεύσουμε τους πολίτες και το περιβάλλον στην Ευρώπη. Μετά την επόμενη συνάντηση θα έρθω να σας αναφέρω και πάλι τα πεπραγμένα μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. Τώρα το λόγο θα πάρουν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Σόνικ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Eksplozja platformy w Zatoce Meksykańskiej to największa tego typu katastrofa. Σας ευχαριστώ πολύ. Η έκρηξη της πλατφόρμας ε, πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικού είναι η πιο σοβαρή καταστροφή 800.000 τόνοι πετρελαίου χύθηκαν στον ωκεανό. 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι καλυμμένα αυτή τη στιγμή από την πετρελαιοκυλίδα. Μεγαλύτερη έκταση από ό,τι δηλαδή ολόκληρε οι κάτω χώρε. Και έχουν χαθεί βέβαια και ανθρώπινε ζωέ, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεδομένης αυτής της καταστροφής, νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε και εμείς ε, τις δικές μας ε, πλατφόρμες εξόριξης στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα πρώτο βήμα για την ε, ασφάλεια στα ευρωπαϊκά ύδατα. Νομίζω ότι αν είχε γίνει στη Βαλτική αυτού του είδους η καταστροφή, τότε η περιβαλλοντική ζημία, η περιβαλλοντική καταστροφή θα ήταν ανεπίστρεπτη, θα ήταν αμετάκλητη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει όλες αυτές οι εξέδρες να παρακολουθούνται, να πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Η ασφάλεια να είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε διεθνή πρότυπα και διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμοστούν στην περίπτωση που προκύψει τέτοιου είδους καταστροφή με δημιουργία πετρελαιοκυλίδας. Επίσης, ε, έχουμε δει αποφάσεις οι οποίες δίνουν ε, άδεια σε κάποιες εξέδρες πετρελαίου και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται πολλές φορές ε, υπό την πίεση των ομάδων πίεσης. Ασκούνται πολιτικές πιέσεις στην Ευρώπη. Είδαμε τι έγινε με το North Stream, τον αγωγό αυτό ε, κατά από τη Βαλτική. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ποτέ 100% ασφάλεια στις πλατφόρμες πετρελαίου που βρίσκονται στους ωκεανούς. Ωστόσο δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε σε λόμπι από τη βιομηχανία να επηρεάζουν τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Από των Σοσιαλιστών Δημοκρατών, ο κ. Σαρσένης έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πολλές φορές απλά αυξάνοντα τα μέτρα πρόληψης, ε, αυτό δεν επαρκεί η πρόσφατη έκρηξη στο κόλπο του Μεξικού έγινε σε μια εξέδρα που είχε κατασκευαστεί μόλις το 2001 και η επακόλουθη βήθησή της προκαλεί μια από τις μεγαλύτερες έως σήμερα οικολογικές καταστροφές. Μέχρι και σήμερα, και έχουν περάσει 29 μέρες από το γεγονός, από το ατύχημα, δεν έχει καταστεί δυνατή η διακοπή της διαρροής. Και όπως είπε και ο κύριος Σόνικ, πάνω από 5.000 τόνοι πετρελαίου εκλείονται στη θάλασσα, σε αυτόν τον κόλπο, κάθε μέρα η τεράστια αυτή ρήπανση συμβαίνει σε μια περίοδο ε, όπου κορυφώνεται η οτοκία πάρα πολλών ειδών πολλών των οποίων είναι υπό εξαφάνιση. Ε, μιλάμε για πέντε ε, από τα, από τα, εφτά είδη θαλάσσιας χελώνας δελφίνια πάρα πολλά κήτη πάρα πολλά σημαντικά θαλάσσια θηλαστικά μοιραία και ο άνθρωπος πλήρωται. Ε, η έκρηξη αυτή, το ατύχημα συνέβη σε μια περιοχή που μόλις ξεκινά να συνέρχεται από τις πληγές που άφησε ο τυφώνας Κατρίνα. Και η ίδια έκρηξη προκάλεσε το θάνατο 11 ανθρώπων. Στην Αμερική όμως λαμβάνουν μέτρα. Το Κογκρέσο ε, το 1981 ψήφισε το μορατόριο που επέβαλε απαγόρευση στην υπεράκτη άντληση πετρελαίου στο 85% της ε, επικράτειας των παράκτων υδάτων της ε, αμερικής. η κυβέρνηση ομπάμα επιβεβαίωσε το μορατόριο μετά το ατύχημα παρά τις αρχικές της αντίθετες δηλώσεις. την ίδια στιγμή όμως στην ευρώπη συνεχίζουν να τίθενται σε λειτουργία πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου κυρίως στη βόρεια θάλασσα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε λειτουργία εκατοντάδε υπεράκτιες πλατφόρμες ε, τόσο για πετρέλαιο όσο και για φυσικό αέριο. Το πρόσφατο ατύχημα στον κόλπο του Μεξικού πραγματικά επιβεβαίωσε το κίνδυνο κυριολεκτικής καταστροφής για το θαλάσσιο περιβάλλον από τις υπεράκτιε εξέδρες άδειας πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναζήτηση και εκμετάλλευση ε, θαλάσσιων αποθεμάτων πετρελαίου εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εβέζου και που αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων ε, σχετιζόμενων με επικίνδυνε ουσίε. Η πρόσφατη καταστροφή μα δείχνει ότι κανεί δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι μια παρόμοια καταστροφή δεν θα μπορούσε να συμβεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καμιά φορά τα μέτρα, απλά αυξάνοντα τα μέτρα πρόληψη, δεν είναι επαρκή. Η κυβέρνηση Ομπάμα μπροστά στο μέγεθο τη καταστροφή αναδιπλώθηκε. Μήπω έχει φτάσει η ώρα πέρα από επιπλέον μέτρα πρόληψης να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ένωση σε ένα ευρωπαϊκό μορατόριο που θα απαγορεύει από εδώ και μπρος την υπεράκτη άδληση πετρελαίου στα της ευρωπαϊκής ένωσης αντίστοιχο με αυτό τον ηπα. επιβάλλεται να δράσουμε άμεσα πραγματικά πριν ένα προαναγγελθέν έγκλημα σε αυτό τον κόλπου του μεξικού χτυπήσει και τη δικιά μας πόρτα. Τώρα για την ε, ομάδα Συμμαχία των Φιλελευθέρων, η κυρία Λεπάζ για τρία λεπτά. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η βήθηση της εξέδρας στις 22 Απριλίου έξω από τις εκθέσεις της Λουιζιάννας ε, προκάλεσε πετρογυλίδα πρωτοφανών διαστάσεων. Τρία ζητήματα τίθονται. Ότι δεν υπάρχει σύστημα πρόληψης τέτοιας διαρροής δεν είναι εύκολο να το καταλάβει κανεί αυτό. Η απουσία επαρκού ελέγχου εκ μέρου των δημοσίων αρχών ε, επί του συστήματος ασφάλειας που υπήρχε και τέθηκε σε εφαρμογή από τους χειριστές τη πλατφόρμας για να αποδειχθεί ο κίνδυνος ρήπανσης και τέλο, ο ειδικό κίνδυνος που σχετίζεται ε, με τη ρήπανση από ε, υδρογονάνθρακες ενό ιδιαίτερα ευαίσθητου περιβάλλοντος. Ο συνάδελφος Σόνικ ε, αναφέρθηκε στην καταστροφή που θα προέγινε κάτι τέτοιο συνέβαινε στην ε, Βαλική θάλασσα. Στην ε, Βόρεια Θάλασσα έγιναν δύο τέτοια επικίνδυνα ατυχήματα. Υπό τις συνθήκες αυτές είναι εντελώς απαραίτητο να προβούμε σε μία έρευνα που θα μας εξασφαλίσει, σε μια μελέτη ε, που θα μας εξασφαλίσει ότι τέτοιου είδους ε, ατυχήματα δεν συμβούν έξω από τις ε, ακτές μας. Τώρα, κύριε Επίτροπε, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε άμεσα ε, για να αποφευθούν τέτοια ατυχήματα στις εξαίρες που βρίσκονται στα δικά μας χωρικά ύδατα ε, και έξω από τις δικές μας ακτές. Ε, τα ελάχιστα μέτρα που αναφέρε αρκετά κύριε Επίτροπε. Δεύτερον, πώς θα φροντίσετε για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων αυτών που δεν πρέπει να μείνουν στο χαρτί και πώς ο έλεγχος της εφαρμογής αυτής θα είναι αποτελεσματικός. Τι έχετε σκοπό να κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση. Τρίτον, ποια είναι τα μέσα που θα εφαρμοστούν για να αποφύγουμε σε περίπτωση ατυχήματο την ρήπαση των ακτών. Γιατί ωραία είναι να έχουμε σκάφη και ε, πολιτοφυλακές και πολιτική άμυνα, ε, αλλά τι ε, συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν. Ε, με, δεν θα είναι απαραίτητο επίσης να, να υπάρχει ένα σύστημα ε, κατανομής των οικονομικών δαπανών και εγγύσεων με σκοπό την αντιμετώπιση των ατυχημάτων αυτών. σε περίπτωση που ε, τίθεται σε κίνδυνο και το θαλάσσιο περιβάλλον ε, και ιδίως τι γνώμη ε, έχετε για την άντληση πετρελαίου σε μεγαλύτερα βάθη και όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Ασένης μήπως ήρθε η στιγμή ενός μορατόριου παράλληλα με αυτό που θέλει να εφαρμόσουν, θέλουν να εφαρμόσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Μήπω έχει έρθει πλέον η στιγμή αυτή. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Τώρα η κυρία Ντουρόν, εκ μέρου τη Συμμαχία των Πρασίνων. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω, κύριε Επίτροπε, ότι θα πρέπει οι μαθητευόμενοι μάγοι στη βιομηχανία να σταματήσουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Διότι υπάρχει δίψα για πετρέλαιο, ε, εκμεταλλεύονται τα πάντα ε, και αυτό σίγουρα πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο ατυχήματο. Οι βιομηχανίε τον τελευταίο καιρό έχουν ε, δώσει μεγαλύτερο βάρο στην εξόρεξη και στην άντληση σε βάρο τη προστασία του περιβάλλοντος. 800.000 λοιπόν τόνοι πετρελίου εδώ και ένα μήνα κάθε μέρα στον ωκεανό καταλήγουν με Τρομερέ καταστροφέ. Έχουμε λοιπόν από τη μια αστρονομικά ποσά για όλο και πιο σε βάθο άντληση και εξόριξη, αντιθέτως όμω πολύ λιγότερα ε, ποσά για την πρόληψη των κινδύνων και την αντιμετώπιση τους. Θα ήθελα και εγώ να πω, όπως συνάδελφοι, διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των εξεδρών. Πετρελαιό να δούμε το επίπεδο ασφάλεια, ε, το κατά πόσο τηρούν τι προδιαγραφέ και επίση να υπάρχει έλεγχο, έλεγχο των εξεδρών ακόμη και αν ε, αυτό ε, γίνεται υπό το, στο, πεδίο, στο πλαίσιο των πεδίων των κρατών μέλων ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πιο εύθραυστα και ευαίσθητα συστήματα. Πήρατε κάποιες πρωτοβουλίε και τις επικροτώ για το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αντίστοιχη τέτοια περίπτωση εφόσον συμβεί στι ακτέ των χωρών μα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρώπη να πάρει και άλλε πρωτοβουλίες για να προστατεύσει ε, μία διαπαντό σε τα πιο εύθραυστα οικοσυστήματα όπω τη Αλλάσκα, παραδείγματο χάρη. Χρειάζεται μία διεθνή σύμβαση όπω ακριβώ αυτή που είναι για την ε, Ανταρκτική. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ε, τηρήσουμε ηγετική στάση σε αυτό το τομέα. Ε, πολύ ε, σημαντικός λοιπόν ο λόγος να επενδύσουμε και στις ανώσιμες πηγές ενέργειας, όπως και για το ηφαίστειο, να μην το αναφέρω το όνομά του γιατί δεν μπορώ και να το πω βέβαια, αλλά επειδή και το ηφαίστειο μας έδωσε κάποια μηνύματα σε ό,τι αφορά τις ε, αέριες μεταφορές, ένα άλλο θέμα είναι και αυτό της εξόρυξης πετρελαίου. Θα πρέπει πλέον να, επιτέλους να καταλάβουμε ότι αυτή η κούρσα για το κέρδος τελικά γυρίζει μπούμεραγκ. Κύριος Τσίτσεστερ τώρα από τους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τη δήλωση του Επιτρόπου. Ο κόσμος έκπληκτος ε, βλέπει να χύνεται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ε, από την εξέδρα που εξεράγει. Και επίσης έχει μείνει έκθαμβος ο κόσμος από την ανικανότητα της βιομηχανίας και των κρατικών αρχών να σταματήσουν τη διαρροή. Ελπίζω ε, να έχουμε θετικές εξελίξεις ε, προσεχώς. Μίλησαν και άλλοι συνάδελφοι ε, για τη Βόρεια Θάλασσα και προηγούμενα επεισόδια, το Piper Alpha στη Βόρεια Θάλασσα. Και Όμω θα πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στα βάθη στα οποία ε, δουλεύουμε στη Βόρεια Θάλασσα από τον κόλπο του Μεξικού, έτσι. Και θα ήθελα να συστήσω προσοχή, προσοχή, μην τρέξουμε τώρα να κάνουμε νέα νομοθεσία. Να είμαστε σίγουροι τι συνέβη να είμαστε σίγουροι αν υπάρχουν κανόνες ε, και θα μπορούσα να το είχαμε προλάβει να συμβεί κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Και επίση να βεβαιωθούμε ότι οποιοδήποτε νέοι κανόνε θα αποτρέψουν τέτοια εξέλιξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν και θεομηνίες και ατυχήματα στη ζωή. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να βεβαιωθούμε και να εγγυηθούμε την πρόληψή του. Και υπάρχει και όριο στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Να σα δώσω και μια τελευταία σκέψη. Όταν σκεφτόμαστε το σχετικό κίνδυνο Τέτοιου είδου ατυχήματα δείχνουν και ποια είναι η σχετική ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας. Έτσι, ας τη δούμε με άλλο μάτι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίζεστερ. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Οαγό για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η διαρροή πετρελαίου στο κόλπο του Μεξικού αποτελεί μια πραγματική οικολογική και οικονομική καταστροφή. Από ό,τι φαίνεται υπήρξαν κάποιες ε, ατασταλίες ε, οι οποίες ε, είχαν διαπιστωθεί όταν το Υπουργείο της, τον δόθηκε άδεια για την εξόριξη Πρόκειται λοιπόν ε, για μια απαράδεκτη και ασυγχώρητη ελαφρότητα που έχει αλόγιστες, ανυπολόγιστες συνέπειες και βλάπτει. Και τη φήμη τον είπα, όταν γνωρίζουμε ότι δίνονται εκατοντάδες ε, άδειες ε, από τα κράτη για τις υπεράκτητες αυτές εξέδρες. Αν αυτές οι άδειες εκχωρούνται με την ίδια ακριβώς ελαφρότητα, νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα για ολόκληρο τον πλανήτη εκλεγμένος από μια υπεραπόμακρη περιφέρεια και από ε, τα υπερπόντια αυτά διαμερίσματα με πάνω από 130 νησιά στις τρεις υπήρους θα πρέπει να πω εδώ ότι πραγματικά ανησυχώ πάρα πολύ για τα νησιά μας ε, λόγω ακριβώς αυτών ε, των ε, έργων ε, εξόριξη πετρελαίου στους ωκεανούς, στις θάλασσες. Γι' αυτό λοιπόν η επιτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα, το καλό παράδειγμα να επανεξετάσει πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφάλειας αλλά και τα προληπτικά προληπτικά μέτρα στις δικές της εξέδρες, ε, υπεράκτες εξέδρες πετρελαίου. Επίσης αυτή η λειτουργική ή τυχαία διαρροή ε, του πετρελαίου ε, στην θάλασσα πολλές φορές οδηγεί ε, στην ιδιωτικοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων τόνων και νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει πρωτοβουλίες ώστε αυτές οι θαλάσσιες εξέδρες ε, να είναι ε, αρμοδιότητα μιας αδιαμφισβήτητης διεθνούς αρχής η οποία ε, θα ασκεί, αν θέλετε, ένα είδος διεθνούς εξής μετά την Κοπενχάγη ε, και προετοιμασία προς το Κανκούν, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα ήταν να ξεκινήσει μια πραγματική παγκόσμια διακυβέρνηση για την έρευνα, για την προστασία και για την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων. Ο κύριος Μάρτιν για ένα λεπτό τους ε, κύριε Επίτροπε, ως ε, γείτονας που μοιραζόμαστε και ε, λίμνες, ε, τη λίμνη Μπόντενζε. Φανταστείτε τι θα, αν γινόταν ε, στην Μπόντενζε, σε αυτή τη λίμνη που έχουμε ανάμεσα στη Γερμανία και στην Αυστρία, αν γινόταν αυτό το πράγμα. Εσείς δεν θα είχατε πόσιμο νερό και εμεί δεν θα είχαμε πια φεστιβάλ το καλοκαίρι. Εντάξει, είναι μακριά οι εξέδρες στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική, άλλοι θα κληθούν να πληρώσουν. Αλλά είστε βέβαιος ότι είμαστε καλά εξοπλισμένοι. Μιλήσατε για καλό συντονισμό. Επανειλημμένα έχουμε δει να μην λειτουργεί ο ασύρματος καν μεταξύ διαφόρων κρατών. Τα έχετε μελετήσει αυτά, τα έχετε ελέγξει. Τι γίνεται με τη νομική κατάσταση, με την νομική βάση. Ε, οι αγωγέ και οι μηνύσει θα ευσταθούν κατά των εταιριών αν συμβεί το κάτι τέτοιο. Και επίση οι ελεγκτικέ αρχές στην Αμερική είδατε πόσο ήταν διαπλεκόμενε με την πετρελοβιομηχανία. Στην Ευρώπη μπορείτε να το αποκλείσετε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρουμε να κάνουμε τα πάντα εκτό από το τάδε. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Αντωνέσκου για δύο λεπτά παρακαλώ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 Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω και εγώ την πρωτοβουλία της Κομισιόν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συζητάμε το θέμα αυτό, έστω και αν το ατύχημα δεν έγινε ε, μέσα στη ζώνη δικαιοδοσίας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών υπάρχουν πολλές πλατφόρμες εκμετάλλευσης πετρελαίου και η δραστηριότητα αυτή θα αυξηθεί εφόσον ε, ο Διεθνή Οργανισμός Ενέργειας διευκρινίσε ότι μόνο 5% των θαλάσσιων κοιτασμάτων πετρελαίου είναι γνωστά αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα είναι τι τι διδάγματα μπορούμε να συναγάγουμε από αυτήν την καταστροφή. Ποια είναι η κατάσταση στα ύδατα όπου υπάρχουν τέτοιου είδου ε, εκμεταλλεύσει ε, στα πλαίσια των κρατών μελών και αν είναι απαραίτητο να ληφθούν επιπλέον μέτρα για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών που εργάζονται σε αυτέ τι εξέδρε, καθώ επίση και μέτρα πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων που έχουν καταστροφικέ συνέπειε. Ένα άλλο δίδαγμα που πρέπει να συναγάγουμε από αυτή την καταστροφή είναι ότι είναι απαραίτητο να εξετάσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το πώς χορηγούνται οι άδειες εκμετάλλευσης αυτών των εξεδρών και ποιες είναι οι πρακτικές που ισχύουν για τις σχετικές συμβάσεις. Πρέπει να ε, είμαστε βέβαιοι ότι θα αναλαμβάνονται πραγματικά οι ευθύνε από τον καθένα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κερδίζουν πάρα πολλά από τέτοιου είδους διαδικασίες και πρέπει να είναι έτοιμες να υποστούν τις συνέπειες αν κάτι δεν πάει καλά. Ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συμβατικές ε, σχέσεις που υπάρχουν ε, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ρίχνουν η μία το βάρος στην άλλη. Δεν πρέπει να ανεχθούμε κάτι τέτοιο στην, εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα μας εξασφαλίζει ότι πραγματικά περιορίζεται ο κίνδυνος επανάληψης ενός τέτοιου ατυχήματος. Η εμπειρία δείχνει ότι τέτοια ατυχήματα οδηγούν σε πολύ σημαντικές ζημιές σε μεγάλες καταστροφές και η Κομισιόν θα πρέπει να εξασφαλίσει ε, ασφαλή εκμετάλλευση του πετρελαίου χωρίς να είναι ιδιαίτερα χαλαρή και να βρει τρόπους να αποτρέψει τέτοιου είδους ε, ατυχήματα. για ένα λεπτό παρακαλώ. Mm, mm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε. Η καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού μας αναγκάζει να ε, εξετάσουμε και πάλι το θέμα των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα ε, να δούμε το θέμα του αγωγού ε, στην Βαλτική θάλασσα που προχώρησε παρά την σύσταση εναντίον που υπήρχε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ποσότητα φυσικού αερίου που θα περάσει από αυτόν τον, από αγωγό ε, σημαίνει ότι θα γίνουν ε, πάρα πολύ εκτεταμένες δραστηριότητες εξόρυξης. Και δεν υπάρχουν ε, αντιλιοστάσια τα οποία θα μπορούσαν να ε, κλείσουν σε περίπτωση ατυχήματος. Αν μπει νερό μέσα στον αγωγό αυτό, ο αγωγός θα καταστρεφόταν παντελώς. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ζητήσω από την Κομισιόν να εξετάσει το είδο των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια επένδυση. Ε, θα πάρουν το λόγο συνάδελφοι για ένα λεπτό ο καθένας, ξεκινώντας από τον κύριο Ρούμπικ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ επίκαιρη η συζήτηση δεν έχουμε λύσει ακόμα τα προβλήματα στον, κόλπο του Μεξικού συγγνώμη, και δεν ξέρω πότε θα εμφανιστούν τα επόμενα και πού. Η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, κύριε Επίτροπε, ε, με το κοινό ερευνητικό κέντρο, με τεχνογνωσία, με άλλα ιδρύματα που έχουμε, έτσι ώστε να περιορίσουμε το συντομότερο από κοινού και αυτή την καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού ή να προσπαθήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μείωση 20% του διοξιδίου του άνθρακα και αντικατάσταση από τις ανανεώσιμες ε, επέλεξε το σωστό δρόμο. Και με την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της εξοικονόμησης μπορούμε πάρα πολλά να πετύχουμε. Εσείς πιστεύετε ότι στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο μπορούμε να συνεργαστούμε με την Νορβηγία, για παράδειγμα, για νέες πρωτοβουλίες. Καντράου έχει το ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και άλλοι προλαλήσαντες ομιλητές, ε, έχω συγκλονιστεί από το γεγονός αυτό ότι ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα επί εβδομάδες να διαραίουν τόσα πολλά βαρέλια πετρέλαιο και να μην μπορούμε να τα σταματήσουμε. Και η BP ε, προσπαθεί όλο και περισσότερο να ε, ελαχιστοποιεί ε, την κατάσταση. Μας κοροϊδεύει, αλλά έχουμε φοβερέ επιπτώσει για το μέλλον και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε εθνικό πλέον, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε στο μέλλον κάτι τέτοιο να είναι αδύνατο. Και από πλευρά διαδικασία και από πλευρά τεχνική να κάνουμε τα συστήματα ασφαλεία έτσι. Βεβαίω έχει και ένα κόστο αυτό. Αλλά το κόστος της απραξίας είναι πολύ ψηλότερο. Στο παρελθόν είχαμε ε, αναλάβει παγκόσμια πρωτοβουλία με ε, το διπλό κήτος στα ε, δεξαμενόπλια και τώρα θα πρέπει να κάνουμε αντίστοιχες προσπάθειες. Ευχαριστώ. Κύριε Καντράουε, το λόγο θα πάρει η κυρία Κάντεμπαχ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Ούτιγκερ, κύριε Επίτροπε, ως μέλος ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και σκιώδη εισηγήτρια για τη βιοπικιλότητα ε, και προσωπικά με έχει συγκλονίσει αυτή η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή ζωής που θα έπρεπε να έχει διατηρηθεί και παρόλη την πρόνοια είπε κάποιο ότι είναι θεομηνίες, τι να κάνουμε, ε, υπάρχουν και ατυχήματα και η δράση μας έχει και όρια. Ναι, αλλά δυστυχήματα δεν έχουμε μόνο στις εξέδρες, έχουμε και σε πυρηνικά εργοστάσια. Διάφορα επεισόδια και ατυχήματα και δυστυχήματα. Ε, ε, και επίσης στην Αυστρία έχουμε μια παραμία που λέει πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει καταστροφή για να ανοίξουμε τα μάτια μας. Να είμαστε δηλαδή επιμηθεί αντί για προμηθεί, Μήπως θα πρέπει να καταλήψουμε και την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και οικονομική και όλη μας την ενέργεια, ε, την πνευματική, για να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες. Ευχαριστώ. Το λόγο ο κύριος Κέλλη τώρα θα πάρει. Ε, Uh, Ευχαριστώ. Σε τελική ανάλυση δεν ξέρω ε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και τι θα συμβεί ε, σε αυτή την περίπτωση ε, και πώς θα αντιδράσουν οι πετρελοβιομηχανίες που έχουν προκαλέσει αυτές τις καταστροφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξίζει συγχαρητηρίων διότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία θα πρέπει να ε, εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα και τους κανονισμούς για να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους καταστροφές ε, στο μέλλον. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και άλλες πηγές ενέργειας, αιωλική, ηλιακή, σε αντίστοιχη περίπτωση, αν δεν τα καταφέρουμε, οι πετρελαϊκές εταιρείες θα συνεχίσουν να ε, κάνουν αυτή την εξόριξη, εξέδρεση όλο και πιο βαθιά στους ωκεανούς, με χειρότερα αποτελέσματα. Thank you, Madam uh, Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η ενεργειακή υποδομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βασίζεται μόνο σε μία προϋπόθεση ότι υπάρχει πλήρης ασφάλεια για την κατασκευή και εκμετάλλευση. Ε, ζητώ κάθε σχέδιο για υποθαλάσσια εξόριξη για μεταφορά υδρογονανθράκων να γίνεται μετά από μία σοβαρή ε, περιβαλλοντική μελέτη. Και τα κράτη-μέλη που έχουν ε, παράκτια ζώνες πρέπει να οργανώσουν ε, ε, μονάδες επέμβασης στην περίπτωση που θα προκύψουν τέτοιου είδους ατυχήματα. Και όλες οι εταιρείες που εξάγουν υδρογονάνθρακες πρέπει να προβλέπεται να πληρώνουν αποζημιώσεις σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ο ολόκληρος ο κόσμος δεν πιστεύει τα μάτια του καθώς παρακολουθεί τα γεγονότα στον κόλπο του Μεξικού. Κανείς δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει ότι μια τόσο μεγάλη και ισχυρή χώρα όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, ότι δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ε, μια τέτοια ε, τραγωδία αποτελεσματικά. Πιστεύω ότι και εδώ στην Ευρώπη επενδύουμε πολύ ε, ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους για να υπάρχουν λύσεις και μηχανισμοί αλλά μερικές φορές η φύση αναλαμβάνει τα ενία. Ε, ποτέ δεν μπορούμε να ε, προβλέψουμε ε, τα πάντα. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σα υπενθυμίσω εγώ μια φορά το Nord Stream. Ε, αν συμβεί οποιοδήποτε τύχημα εκεί πέρα, εμεί θα είμαστε υπεύθυνοι. Πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά ακόμη μια φορά. Να συζητήσουμε το θέμα τη ασφαλού εκμετάλλευση του Nord Stream. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια. Σου ο Σέτιγκερ. You have the floor, Mr. Commissioner. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, και εγώ έχω συγκλονιστεί όπως και εσείς. Όχι μόνο υπό την ιδιότητά μου ω Επιτρόπου, αλλά και ω πολίτη. Γιατί εδώ βλέπουμε πώς καταστρέφεται η φύση για χρόνια ολόκληρη και, πώς ε, παρενοχλείται στη λειτουργία του το σύστημα, το οικοσύστημα. Ωστόσο, ψυχραιμία το άγχος, η ιστερία, η αγωνία θα ήταν λάθος. Ακόμα δεν ξέρουμε καν τον ακριβή λόγο της ε, έκρηξης. Η τεχνολογία ήταν ανθρώπινο σφάλμα. Δεν ξέρουμε ποιος έσφαλε. Εγώ εμπιστεύομαι και την Αμερικανική κυβέρνηση και την κοινή γνώμη ότι θα το διερευνήσουν με την ίδια μεθοδικότητα και την ίδια επιμέλεια ε, που ακολουθούμε και εμείς στην Ευρώπη σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης πιστεύω ότι ο πληθυσμός των ΗΠΑ της Αμερικής είναι επίσης συγκλονισμένο και περιμένει την ίδια μεθοδικότητα και συστηματικότητα στην εξέταση. Γι' αυτό λέγω λοιπόν ότι εμπιστεύομαι αυτή τη βιομηχανική χώρα, την Αμερική, και την τεχνολογία της και τις τεχνικές της δυνατότητες και τη δημοκρατία της. Δεύτερον, θα πρέπει να αρχίσουμε να εγκαταλείπουμε σιγά σιγά το πετρέλαιο. Αλλά ε, τι τελευταίε δεκαετίε γενιέ ολόκληρε οι βιομηχανικέ χώρε έχουν πάρει το δρόμο του πετρελαίου. Έχουν ακολουθήσει αυτή την οδό και οι πολίτε μα. Έχουν πάνω από 200 εκατομμύρια γιοταχή στην Ευρώπη. Και εσείς και εγώ. Ταξιδεύουμε πολύ. Και εγώ και μάλιστα πετάω και πολύ για λόγου υπηρεσιακού. Το Σαββατοκύριακο εκατοντάδες χιλιάδε ε, θα πάνε ε, στη Μαγιόρκα για τις διακοπές της Πεντηκοστής. Και για την Ισπανία και την Ελλάδα ακούμε ότι μόνο ο τουρισμός μπορεί να μας σώσει από την κρίση. Άρα περισσότερες πτήσεις για Αθήνα, για Πάλμα, για Μαρμπέγια και πάει λέγοντας. Εμείς λοιπόν όλοι μας καταναλώνουμε πετρέλαιο και εσείς και εγώ. Γιατί φαίνεται ότι ακόμα και αυτό το κοινοβούλιο δεν έχει χτιστεί ε, ενεργειακά με ε, ε, τρόπο εξοικονόμησης. Έχουμε, ας πούμε, περισσότερα φώτα από βουλευτές εδώ σήμερα. Και θα πρέπει σιγά σιγά να καταλείπουμε το δρόμο του πετρελαίου. 20% ε, πηγές ενέργειας σε 20 χρόνια. Ήδη προετοιμάζουμε ένα οδικό χάρτη για το 2050 και κατά τη διάρκεια του έτους θα σας δώσουμε τις διάφορες εναλλακτικέ προτάσεις. Αυτά τα βλέπουμε από μελέτες ότι σε τέσσερις δεκαετίες μέχρι 80% της ε, ενέργειας που χρειαζόμαστε θα πρέπει να προέρχεται από άλλες ενέργειες, μη ορυκτές μορφές και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και να ξεφύγουμε από το πετρέλαιο. Έχουμε ευκαιρία, αλλά ε, τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα δεν είναι το παρόντος ακόμα, ούτε, ούτε το αύριο καν δεν είναι. Και χρειαζόμαστε και πετρέλαιο και βενζίνη για αρκετά χρόνια ακόμα. Ποιο είναι το γεγονό τώρα και τι είναι σαφές ότι όποιο ε, ψάχνει πετρέλαιο και κάνει εξόριξη στο ε, κόλπο του Μεξικού ε, και στη Βόρεια Θάλασσα Το κάνει για να μειώσει την εξάρτησή του από το πετρέλαιο. Γιατί αν δεν ψάχναμε εμεί και δεν είχαμε δική μα προσπάθεια, θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από χώρε πετροπαραγωγέ που δεν είναι πάντα οι δημοκρατικότερε. Και υπάρχει μια σημαντική διαφορά. 150 μέτρα βάθο είναι ε, στη Βόρεια Θάλασσα, ε, μέχρι 200 μέτρα. Στον κόλπο του Μεξικού είναι 3.000 μέτρα. Μέχρι και 4.000 μέτρα ο βυθός. Με όλα τα συμπαραμαντούντα και τις ε, δυσκολίες να εξασφαλιστεί η παραγωγή. Λοιπόν, 150-200 μέτρα φτάνει κανείς με επανδρομένα υποβρύχια. Ενώ στον κόλπο του Μεξικού στις 3.000 μέτρα είναι πάρα πολύ βαθιά για να φτάσει ο άνθρωπος πάρα πολύ βαθιά για να έχουμε ε, τεχνική ασφάλεια. Εγώ εμπιστεύομαι επίσης και τα κράτη-μέλη μας. Έχουμε κάθε λόγο να εμπιστευόμαστε τις εθνικές μας αρχές, τους οργανισμούς και τους τεχνικούς μας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Νορβηγίας, της Δανίας, ότι ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνουν. Και στην εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΜΣΑ, τον οργανισμό μας ε, συνεργάζονται ε, με τις εθνικές υπηρεσίες και έχουμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και συνεργασία για την ασφάλεια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών που βρέχονται από θάλασσες. Βεβαίως, έχουμε και τον North Stream και χρειάστηκε να ελέγξουμε και εκεί την ασφάλεια. Ήταν περίπλοκα τα ζητήματα ε, της αδειοδότησης για την ασφάλεια, ε, φτάσανε σε όλα τα στάνταρ και πρέπει να σας πω ότι το Nord Stream είναι πιθανότατα η πιο σύγχρονη μορφή αγωγού και η πιο ασφαλής μορφή αγωγού φυσικού αερίου στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. Υπάρχουν και διαφορές αν υπάρχει ένα πρόβλημα στο φυσικό αέριο, μπορεί να κλείσει τη στρόφιγγα στην πηγή ή στην ακτή. Δεν μπορεί να συγκριθεί το Nord Stream μετά όσα συνέβησαν στον κόλπο του Μεξικού. Και τελικά, θα πρέπει, σας είπα, να πάρουμε το δρόμο που εγκαταλείπει το πετρέλαιο, αλλά αυτό θα χρειαστεί δεκαετίες. Ο καθένας από εμά και στην πολιτική και στην κοινωνία θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει, να αρχίσουμε να, να απαγκιστρωνόμαστε από το πετρελαίο και στο μεταξύ να ελέγξουμε τα στάνταρ, τις προδιαγραφές, ε, τις οδηγίες, τους νόμους και ό,τι άλλο θέλετε σε υψηλότατο επίπεδο. Έχουμε κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Τις απαντήσεις θα τις έχουμε το φθινόπωρο και τα στοιχεία και όταν θα ε, έχουμε κάνει αυτές τις σκληρές ερωτήσεις με τα ερωτηματολόγια στις εταιρείε, θα σας αναφέρουμε τις απαντήσεις και πιστεύω ότι οι εταιρείε που ασχολούνται με την ενέργεια τα έχουν καταλάβει αυτά. Και υπάρχουν και ζητήματα αστικής ευθύνης για την αποζημίωση. Ήδη υπάρχουν αυτά. Κατά τα άλλα, στις Ηνωμένε Πολιτείε δεν αμφισβητεί κανένας ενεχόμενος ε, για το ποιος φταίει και ποιο, ότι πρέπει να πληρώσει και αυτός που φταίει. Και σήμερα σας λέγω ότι αυτό είναι της τάξης των δισεκατομμυρίων. Και στην Ευρώπη έχουμε ε, ζητήματα περιβαλλοντικά και αστικής ευθύνης που ρυθμίζονται. Ο Ριπένον πληρώνει και τα λοιπά. Αυτά είναι γνωστά. Και ε, σίγουρα ε, αυτό θα ενισχύσει και την προφύλαξη και την πρόληψη. Σε λίγες εβδομάδες λοιπόν θεωρώ ότι θα γνωρίζουμε ε, αν χρειάζεται νέα νομοθεσία ή νέα τεχνολογία και θα ξανάρθουμε να σας ενημερώσουμε. Ε, οι τοποθετήσεις σας δείχνουν πόσο σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα πέρα από πολιτικές ομάδες και κόμματα και ε, θα πρέπει να είμαστε εδώ πραγματικά ε, με πρόληψη και εμφροφύλαξη και όχι να ερχόμαστε εκ των υστέρων να λύνουμε τα προβλήματα. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έλξε κυρίε και κύριοι συνάδελφοι εδώ. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάρκειας.